όπως επίσης και τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα θεωρία, ότι δεν είναι παρόντες όλοι οι βουλευτές στην Ολομέλεια. Υπάρχουν πολλές απουσίες λόγω μιας ε, τεχνικής βλάβης η οποία έχει μπλοκάρει όλα τα αεροδρόμια στο Βέλγιο Ελπίζουμε να μπορέσουν να ανοίξουν τα αεροδρόμια αυτά στις 4 το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα. Είναι σωστό αυτό για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και να είναι πληροφορημένοι οι βουλευτές που παρακολουθούν. Λοιπόν, τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 21ης Μαΐου είναι στη διάθεση των βουλευτών.